Przewodniczący! Uh, ah, αγαπητοί συναδελφοί, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Wznawiam sesję. Otwieram Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση που διακόπη στις 17 Ιουνίου 2010. Τα πρακτικά της συνεδρίας